Now, uh, Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Ξεκινάμε με την έκθεση της κυρίας Ντελβό για την πρόθεση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων. Έχουμε λίγους ομιλητές. Ο κύριος Τζαμπάσκι. Παρακαλώ.